Uh, colleagues, uh, good afternoon. Um, Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Καθότι δεν είναι παρόν σήμερα ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δεν θα είναι ε, στη διάθεσή μας καθ' τη διάρκεια της ε, συνεδρίασης ε, και καθότι βρίσκεται... και μου ζητήθηκε να προεδρεύσω σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω αυτό να μην οδηγήσει σε πολλές διαμαρτυρίες. Ε, οι οι συγητές λοιπόν ζήτησαν τις εξής ε, αλλαγές στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα. Καταρχήν, το σημείο 4 για την ποινική προστασία του ευρώ και των άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη ε, την, η έκθεση της κυρίας Μάκιντα δηλαδή θα συζητηθεί στις 4 και 4 περίπου. Και αυτό είναι ο λόγος που θα ξεκινήσουμε με το σημείο 5 ε, την απόφαση του δικαστηρίου και το σημείο 6 την αντιπροσωπεία ΛΥΜΕ ε, ε, στον οργανισμό EU-LISA. Κατόπιν της, της εισηγήτριας η συζήτηση της γνωμοδότησης και της θα, θα αναβληθεί. Ε, το σημείο 15 στη μέση διαταξή σας, η ψηφοφορία Γκάμπριελ, θα ε, αναβληθεί σε προσεχή συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ με τις ε, τροποποιήσεις αυτές λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, θα ήθελα να υιοθετήσουμε την ημέρηση διάταξη. ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ να εγκρίνετε τις συστάσεις των συντονιστών. Καταρχήν, ορισμός εισηγητού. Και βλέπω με μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετή ικανοποίηση ότι έχω οριστεί εισηγητής της γνωμοδότησης της 29ης ετήσιας έκθεσης για παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του ε, Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το 2011. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Σημείο 3. Η τρέχουσα κατάσταση των ενεξελίξεων διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Ε, τριμερής διάλογος για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος μα, ο κύριος ε, Λοπέζη Κίγια, προείδρευσε σε δύο ε, τριμερείς διαλόγους για να βρεθεί λύση στο θέμα των κατεξοδότηση πράξεων και τον προγραμματισμό εντός των ε, ε, δημοσιονομικών προγραμμάτων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΛΥΜΠΕ. Εμείς από πλευρά του Κοινοβουλίου έχουμε εργαστεί πάνω σε μια συμβαστική πρόταση που θα πληρεί τις προϋποθέσεις της διάσκεψης των Πρόεδρων και των συντονιστών μας και βασίζεται σε προηγούμενα άλλων διαπραγματεύσεων σε άλλες επιτροπές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ε, στα θέματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη. Η Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο, ε, δεσμεύτηκε να ε, διαβιβάσει γραπτό τι προτάσει τη. Ζητήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση να μα δώσει τι προτάσει τη το αργότερο Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν έχει συμβεί. Ο Πρόεδρος ε, φυσικά μαζί με όλους τους ε, συζητητές ε, ε, θα συνεχίσει να υπερασπίσετε τα προνόμια του Κοινοβουλίου στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Θα σα κρατήσουμε ενήμερου για οποιασδήποτε νέε εξελίξει. Και για τι εξελίξει μετά την παραλαβή τη ανακοίνωση αυτή τη Κομισιόν. Περαιτέρω τριμερή διάλογο μπορεί να πραγματοποιηθεί στι 25 Σεπτεμβρίου. Ο Πρόεδρος επίσης θα ε, υποβάλει αναφορά στον πρόεδρο Σούλτσε που θα κάνει τριμερή διάλογο ε, υψηλού επίπεδου ε, κατά τι προσεχείς εβδομάδες. Συνάδελφοι, προχωρώ τώρα στο σημείο 5 την απόφαση στην, υπόθεση 648 11 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το υπεύθυνο κράτο μέλος για την εξέταση αιτήσεω ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου που υπέβαλε αιτήσει και σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι το κράτο στο οποίο βρίσκεται ο λόγο ανήλικος μετά την υποβολή αυτό αιτήσεω ασύλου. Συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στη νομική υπηρεσία για να μας παρουσιάσει αυτή την υπόθεση. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο η υπόθεση αυτή, καθότι σε κοινή πολιτική δήλωση που έχει επισυνευθεί στην αναδιατύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου, ε, ε, ε, ελήφθη αυτή η απόφαση και έχει δεσμευτεί η Κομισιόν ε, να σχεδιάσει μια νέα νομοθετική πρόταση με προσαρμογή του κειμένου του κανονισμού του Δουβλίνου. Εάν η υπόθεση του δικαστηρίου αλλάξει τον κανονισμό, τότε η εν λόγω διάταξη σχετίζεται με ασυνόδευτους ανήλικους που κάνουν αίτηση για διεθνή προστασία. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην νομική υπηρεσία να μας κάνει μια παρουσίαση. Παρακαλώ. Η περίπτωση στην οποία αναφερθεί αφορά την προσαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. Ξέρετε ότι η αναθεώρηση ήταν τμήμα του πακέτου η αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας Ξέρετε ότι αναφέρεται ο κανονισμός αυτός στον καθορισμό των κριτηρίων του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας υποψηφιότητας ασύλου έτσι ώστε η διαδικασία να γίνεται μόνο σε ένα κάθε ένα μέλος κάθε φορά. Υπάρχει μια ιεραρχία θα έλεγα για τις αιτίε και τους λόγους για τους οποίους είτε θετικά είτε αρνητικά ορίζεται ένα κράτος μέλος ως υπεύθυνο. Σε αυτή την περίπτωση είναι η χώρα πρώτης αίτηση που είναι υπεύθυνη. Μπορεί να ληφθεί επίσης πρωτοβουλία ανεξάρτητα επί τη βάση της λεγόμενης αρχής της κυριαρχίας. Παρέχονται επίσης οι κανόνες επί τη βάση των οποίων οι πολίτες τρίτων χωρών καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσει τους σε άλλη χώρα από τη χώρα στην οποία έχουν μεταφερθεί και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται οι διαδικασίες μεταφοράς των αιτήσεων στην επόμενη χώρα. Η διαδικασία ξεκίνησε με αίτημα προκαταρκτικής λήψης απόφασης από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου, συγκεκριμένα από το εφετείο της, ε, ε, ε, της συγκεκριμένης χώρας επί τη βάση του καθορισμού της χώρας που είναι υπεύθυνη για την ε, εξέταση της υποβολής ε, αιτήσεως ασύλου για χορήγηση ασύλου για, ε, για ανηλίκους. Υπήρχαν δύο περιπτώσεις παιδιών από την Ερυθρέα και ένας από το Ιράκ δεν υπήρχαν χώρες της οικογένεια σε άλλες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχαν συγγενείς, συγγνώμη, των παιδιών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση είχαν κατατεθεί αιτήσει και στην Ολλανδία και στην Αγγλία και στην Ιταλία και αποφασίστηκε οι ανήλικοι να μεταφερθούν στις χώρες αυτές που θεωρούνται υπεύθυνοι για την εξέταση ε, της αιτήσεω τους. Οι ανήλικοι αυτοί αμφισβήτησαν την ομιμότητα της μεταφοράς τους πριν από την απόφαση για τη μεταφορά των δύο ανηλίκων και μετά από την μεταφορά ενός από τους ανηλίκους αποφάσισαν επί τη βάση της ρήτρας κυριαρχίας ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να προχωρήσουν στην εξέταση της αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της, αυτής της συμφωνίας του Δουβλίνου. Τι προβλέπει το 6. Πρώτον, το εάν ένας ανήλικος έχει συγγενείς σε μία χώρα μέλος. Αυτό εξετάζεται πρώτο. Σε αυτή την περίπτωση, το συγκεκριμένο περίπτωση μάλλον η χώρα είναι η υπεύθυνη προς το συμφέρον φυσικά του παιδιού, του ανηλίκου. Όπως είπα οι τρεις ανήλικοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαν συγγενείς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα μέλος όπου ο ανήλικος κατέθεσε την αίτησή του πρώτον, κατά πρώτον είναι υπεύθυνη. Τι γίνεται όμως αν ο ανήλικος έχει καταθέσει αίτηση σε πάνω από μία χώρα, όπως ακριβώς οι τρεις αυτοί ανήλικοι. Σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 6 δεν προβλέπει μία λύση για τέτοια απόφαση. Όπως ενθυμίστε το άρθρο 6 ήταν ένα από τα βασικά θέματα διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λόγω της έλλειψης συγκεκριμένης ρύθμισης για τις περιπτώσεις πολλαπλών αιτήσεων. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά πρώτα να μιλήσω για την απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο είπε ότι στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ένας μη συνοδευόμενος ανήλικος χωρίς συγγενείς σε μια χώρα, που έχει καταθέσει αιτήσει για χορήγηση ασύλου σε πολλές χώρες, τότε η χώρα στην οποία είναι παρόν ο ανήλικος όταν κατέθεσε την αίτησή του είναι αυτόματα υπεύθυνη. Για να καταλήξει στην απόφαση αυτή το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ακριβώς το περιεχόμενο των ισχυουσών ρυθμίσεων και δεν καθορίζει το είδος της αιτήσεως ε, ε, και τον χρόνο υποβολής της. Ε, δεν θεωρείται ότι η πρώτη κάθε φορά ε, ε, αίτηση είναι αυτή που καθορίζει τη χώρα. Μάλιστα, όπως είπε ο Γενικός Εισαγγελέας στην δική του νομοδότηση, το άρθρο 6 θα πρέπει να θεωρηθεί σαν η μοναδική νομική ρύθμιση για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Δεύτερον, το δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 6 επί τη βάση των στόχων του κανονισμού, την αποτελεσματική και άμεση χρήση των διαθεσίμων διαδικασιών και των προβλέψεων του άρθρου 6 πιο συγκεκριμένα, που έχουν σαν στόχο ακριβώς την κάλυψη των αναγκών των ασυνοδεύτων ανηλίκων. Καθόρισε το δικαστήριο ότι οι προβλέψεις ισχύουσες για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, που είναι ένα σημαντικό τμήμα ε, του θέματος της διεθνούς προστασίας. Είπε το δικαστήριο ότι η διαδικασία για τον καθορισμό του υπεύθυνου κράτους, της υπεύθυνη χώρας μέλους, δεν θα πρέπει να κρατά πολύ και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αδικαιολόγητες μεταφορές. Επί τη βάση του 15 του κανονισμού του Δουβλίνου, το δικαστήριο προχώρησε ε, στην ε, ερμηνεία της συγκεκριμένης ρύθμισης. Κατέληξε ότι η ερμηνεία αυτή στηρίζει τις προηγούμενες αποφάσεις επί τη βάση της προστασίας των συμφερόντων του ανηλίκου. Και γι' αυτό η πρόβλεψη θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι καθορίζει πράγματι ως υπεύθυνο κράτος μέλος, το κράτος μέλος το οποίο είναι παρόν ο ανήλικος όταν καταθέτει την αίτηση. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ζήτησαν κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με το προηγούμενο άρθρο 6, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί στα πλαίσια της αναθεώρησης σε άρθρο 8 και καθορίζει όπως είπα την υπεύθυνη χώρα μέλος αντρεφερέντουμ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης και το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να υπάρξει μεγαλύτερη καθαρότητα σε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 6 έως 6 νυν 8 έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες μετακινήσεις ανηλίκων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο δεν ήταν σύμφωνο και είπε ότι δημιουργείται ε, ο κίνδυνος θα έλεγε κανείς του shopping σε, ε, σε σχέση με τις καταθέσεις αιτήσεων για χορήγηση ασύλου και η διαδικασία αυτή από το Συμβούλιο θεωρήθηκε απρόβλεπτη και με πιθανώς κακές συνέπειες. Έτσι λοιπόν επί τη βάση του 6α γίνεται αναφορά στην χώρα στην οποία κατέθεσε ο ανήλικος την αίτησή του χωρίς να υπάρχει αναφορά σε πολλαπλές άλλες αιτήσει ακριβώς για να προστατευτούν τα συμφέροντα του ανηλίκου. Συμφωνήθηκε επίσης με μέσο μιας κοινή δηλώσεως η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης μαζί με τον κανονισμό Δουβλίνο 2 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην αναθεώρηση των ρυθμίσεων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους επί τη βάση της φάσης 6C 648 του 2, μέχρι, ε, το, μέχρι το τέλος του 2000, ε, μέχρι τον Ιούλιο μάλλον του 2016 για την καλύτερη προστασία του ανηλίκου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρούσα φάση αναλύει το περιεχόμενο αυτής της απόφασης και η απόφαση αυτή είναι σημαντική για την ερμηνεία του άρθρου 8 του νέου κανονισμού του Δουβλίνου αυτή τη στιγμή θεωρηθεί ότι είναι εφαρμόσιμος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένας-δυο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα έλεγα να τους ακούσουμε και μετά θα στραφώ στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ράγεν. Πρώτα απ' όλα η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να παραδεχτώ ότι σε αυτή την Επιτροπή, στο σώμα μας, δεν συγκινείται κανεί συχνά τόσο, σε τόσο προσωπικό επίπεδο από τα λόγια τη νομική υπηρεσία. Σήμερα φτάσαμε ακριβώ σε μια τέτοια στιγμή. Έτσι αισθάνομαι. Και να θυμίσω σε εσά, Πρόεδρε, και στου υπόλοιπου Σκιώδη για αυτό το θέμα, ότι αγωνιστήκαμε. Αγωνιστήκαμε και προσπαθήσαμε σκληρά έω το τέρμα. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τους υπόλοιπους κοιόδης, είτε είναι παρόντε είτε όχι, για αυτά που πετύχαμε. Κάποιες φορές μπορούν να γίνουν και θαύματα. Όπως όλοι ξέρουν, ε, εγκρίναμε ένα κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου τον Ιούνιο. Και ο κανονισμό του 3 αποτελεί μέρο αυτού του συστήματο. Και για αυτόν τον κανονισμό είμαι εγώ εισηγήτρια. Ένα από τα πιο ακαθόδη ζητήματα, προκειμένου να καταλήξουμε σε τελική συμφωνία και μετά από πολλά εμπόδια που είχαμε να επερπηδήσουμε, ήταν ακριβώ το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων και το πού θα πρέπει να εξετάζεται η αίτηση ασύλου. Ο προηγούμενο κανονισμό Δουβλίνου έλεγε ότι πρέπει να γίνεται στη χώρα, παραθέτω, όπου οι αιτήσει ε, υποβάλλονται. Αυτό είχε ερμηνευτεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως ε, επιταγή για αναπομπή του ανεασυνοδευτών υλίκου στην πρώτη χώρα εισόδου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μας θέλουν να το διευκρινίσουν αυτό προσθέτοντα ότι θα πρέπει να είναι η προσπατότερη αίτηση που λαμβάνεται υπόψη. Το Συμβούλιο ήθελε και αυτό να το αποσαφηνίσει, αλλά επιπλέον να προχωρήσει ώστε η πρώτη αίτηση να λαμβάνεται υπόψη. Ήταν αδύνατο λοιπόν να βρεθεί συμβαστική λύση μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το θέμα αυτό. Τέλος, ε, καταλήξαμε στη συμφωνία να παραμείνουμε πιστοί στο κείμενο του προηγούμενου κανονισμού, συμπληρώνοντα το εξή. Ε, αρκεί να είναι όλα αυτά προς το μεγαλύτερο έοφυλο του ασυνόδευτου ανηλίκου. Και μετά έγινε και μια δήλωση με αναφορά στην δικαστική αυτή υπόθεση που μόλις μας ε, διάβασε η Καμίλα τις λεπτομέρειές της. Η κοινή δήλωση λοιπόν όλων των θεσμικών οργάνων λέει ότι αφόσον υπάρξει απόφαση δικαστηρίου για το θέμα αυτό, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου προκειμένου να το ευθυγραμμίσει με την απόφαση του δικαστηρίου. Χαίρομαι πολύ που είδα το πόρισμα αυτό από την ε, δίκη ε, στο δικαστήριο, διότι αυτό αποδεικνύει ότι η ερμηνεία μας ήταν σωστή. Οι ανήλικοι δεν πρόκειται να μετακινούνται ε, από μια χώρα σε μια άλλη αυτής τη Υπήρου θα πρέπει να αποζητούμε την σταθερότητά τους και ακριβώς να εξετάζει τη διατησή τους στην χώρα όπου είναι και παρόντες σωματικά. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς έχει γίνει αντιληπτή η απόφαση αυτή στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι για μένα είναι σαφές το τι σημαίνει. Θα πρέπει να υλοποιηθεί ως έχει. Ο ασυνόδευτος ανήλικος θα πρέπει να μην υπόκειται σε ταλαιπωρίε και μετακινήσει βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου. Θα ήθελα να μα διαφωτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν αυτό ή όχι έχει γίνει σεβαστό τώρα και αν ε, έχει τηρηθεί από τα κράτη-μέλη. Θεωρώ δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της δικαστικής απόφασης θα ε, επιστρέψει στο Κοινοβούλιο προτείνοντας αναθεώρηση του άρθρου 8.4 προκειμένου να ευθυγραμμιστεί αυτό με το νέο κανονισμό του Δουβλίνου και με την ε, πρόσφατη δικαστική απόφαση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή και εξάστερη. Πότε θα γίνει αυτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Με αυτά κλείνω και σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονώ να ακούσω την απάντηση. Βεβαίω, θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευκαιρία να απαντήσει σε συγκεκριμένε ερωτήσει όπω αυτή προ το τέλο. Τώρα να αποτίσω φορό τιμή σε εσά, κυρία Βίξτρομ, για τη δουλειά σα. Συγχαρητήρια για όλο σα το έργο στον τομέα αυτό και με άλλου και με τον Μάρκομ Χάρμπορ και άλλου συναδέλφου. Θα ακούσουμε τι θα πούν σήμερα το απόγευμα στι παρεμβάσει του. Μετά η κυρία Σίπολ. Ja, vielen Dank. Ich kann Ευχαριστώ πολύ. Μετά από την συνάδελφο Βίκστρομ, νομίζω ότι μπορώ να είμαι αρκετά σύντομη. Ε, ιδιαίτερα με απασχολεί το εξής. Μια απόφαση είναι ένα πράγμα, αλλά οι συνέπειες στην πράξη είναι άλλες. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τι συνέπειες θα υπάρχουν από αυτήν την απόφαση και στο θέμα του δικαίου του ασύλου από τη μία και το πώς ε, θα χειριστούμε τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους ε, από την άλλη. Είναι θέματα που θα οδηγήσουν σε διάφορες συζητήσεις και προσωπικά θα ήθελα να πω ότι είτε με την παλιά διατύπωση είτε με τη νέα ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικός διότι οδηγεί ε, όχι σε ε, δίκαιη κατανομή ε, των, ε, των ασύλων σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους θα δούμε τώρα μία νέα πρακτική που βασίζεται περισσότερο στις ανάγκες των ανηλίκων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μορδάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά, διότι νομίζω ότι αυτό το θέμα αφορά ιδιαίτερα στη χώρα μου, την Ουγγαρία. Έχουμε όλο και περισσότερους ετούντες άσυλο που περνούν στη χώρα και αυτό έχει προκαλέσει εντάσεις πρόσφατα. Κυρίως γιατί υπάρχει ένα νέο καταβλισμός για τους ετούντε άσυλο στο Πέτσεν στην ε, Ουγγαρία. Επειδή εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ε, εγκαταλείπουν τις χώρες τους λόγω της, των άδικων ευθοπραξιών και της ε, παράλογης τάσης του δυτικού κόσμου αυτό ε, πιο πολύ καταδεικνύει την ε, ε, έλλειψη ισορροπίας στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό. Είναι κακό και για αυτούς ανθρώπους, τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και για όσους ε, πρέπει να υποφέρουν από τις κοινωνικές εντάσεις στη χώρα ε, υποδοχής. Δεν θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά να είναι αντικείμενο συζήτηση. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμη δεν καταλαβαίνω ε, τι συμβαίνει, γιατί συζητούμε την έννοια του ασυνόδευτου ανηλίκου που είναι και ε, το Νάσιλο. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, πώς γίνεται, πώς φτάνει ένα τέτοιο παιδί στην Ευρώπη. Βεβαίω δεν μπορεί ένα δεκάχρονο ξαφνικά από τον τρίτο κόσμο ένα πρωί να ξυπνήσει και να, να αποφασίσει να βρεθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα για να ζητήσει άσυλο. Μήπω λοιπόν εδώ μιλάμε για διακίνηση ανθρώπων, για εμπορία ανθρώπων, μήπω αυτό υποκρύπτεται πίσω από το θέμα που συζητάμε, γιατί έχουν γίνει τεράστιε έρευνε για το θέμα αυτό και θα έπρεπε να συνεχιστούν. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ την εκπροσώπη τη νομική υπηρεσία για την παρουσία τη, αλλά Το θέμα είναι πώς θα ερμηνεύσουμε εμείς τη δικαστική απόφαση για τις αιτήσει των ανηλίκων. Η πρώτη αρχή στην οποία πρέπει να παραμείνουμε πιστό είναι το, πιστή είναι το συμφέρον του παιδιού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το, το, το, το σημαντικότερο συμφέρον ε, και όφελο του παιδιού που να προστατεύσουμε είναι το να μεγαλώσει στη χώρα στην οποία γεννήθηκε, να μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του και να ζει στον πολιτισμό από τον οποίο προέρχεται. Ε, τώρα στην Ευρώπη, παιδιά από τον τρίτο κόσμο, γιατί πρέπει να γίνονται δεκτά. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι ο τρίτο κόσμο δεν είναι ένα μέρο που θα πρέπει να ζουν ε, παιδιά. Έτσι ενθαρρύνουμε του εμπόρου να εμπορεύονται και παιδιά. Um, θα πρέπει να θέσουμε το θέμα στη σωστή του προοπτική. Αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα το απόγευμα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Εμείς δεν συζητάμε το σύνολο του θέματος των ασυνόδευτων ανηλίκων γενικότερα, διότι αυτό είναι μια ευρύτερη συζήτηση και γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε το θέμα στα πλαίσια της αποφάσεως που έγινε δεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους ανηλίκους, τους ασυνόδευτους την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και αναφέρομαι στην έκθεση Γκρισμπέκ και στις προσπάθειες οι οποίες γίνονται παράλληλα για να εντεπιστούν οι ενήλικοι οι οποίοι προχαρούν σε πρακτικές τράφικινγκ, σωματεμπορίας και που θέτουν τους ανήλικους σε τέτοια κατάσταση. Είναι ένα παράλληλο θέμα αυτό. Εμείς λοιπόν ζητάμε, συζητάμε σήμερα ένα κομμάτι του θέματος της αντιμετώπισης των ανηλίκων και η ανάμειξη ανάμεσα στις ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις και την απόφαση του δικαστηρίου δείχνουν ότι απαιτείται μια υποκειμενικότητα ε, στην περίπτωση της σωστής αντιμετώπισης αυτών των ανηλίκων. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς σε επίπεδο νομικό, αλλά απαιτείται να υπάρξει η μέγιστη δυνατή καθαρότητα και απλότητα στις αποφάσεις αυτές. Ακριβώς επειδή μιλάμε για τη συγκεκριμένη κατηγορία των ανθρώπων ανεξαρτήτως των συνθήκων που τους οδήγησαν εκεί και απαιτείται η μέγιστη ευρύτητα πνεύματος. Στρέφομαι τώρα παρακαλώ την Ευρωπαϊκή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναφερθεί στα φαρμοστικά θέματα. Ο κύριος Στίβεν Ράιαν έχει τον λόγο αναπληρωτής υπεύθυνος τμήματάρχης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την απόφαση αυτή και η Επίτροπος Μάλστρομ νομίζω το ανέφερε αυτό ε, στην ε, Ολομέλεια όταν υιοθετήθηκε το πακέτο ασύλου. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η απόφαση αυτή. Επιβεβαιώνει τις απόψεις ε, της Κομισιόν σχετικά με την ερμηνεία του, παρόντος, ε, του ισχύοντος κανονισμού του Δουβλίνου. Η διατύπωση παραμένει ως έχει, αλλά τώρα έχει διευκρινιστεί η ουσία και επιβεβαιώνει ότι οι περιττές μετακινήσεις παιδιών μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει να αποφεύγονται και ότι η αίτηση του παιδιού θα πρέπει να εξετάζεται στο κράτος μέλος όπου είναι παρόν το παιδί ε, για να προστατευτούν ε, τα συμφέροντά του. Ε, και στην κοινή δήλωση μας τα λέμε αυτά που έγινε όταν υιοθετήθηκε η απόφαση, θα πρέπει να εξετάσουμε αν θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί το άρθρο 8.4. Εάν είναι να υπάρξει τροποποίηση, θα πρέπει να είναι ε, στοχευμένη στην ε, συγκεκριμένη διάταξη. Η Κομισιόν ακόμα εξετάζει εσωτερικά το εάν θα είναι απαραίτητη μια τέτοια τροποποίηση. Μία τροποποίηση που θα διευκρινίζει ε, το νόημα της ε, θα είναι ε, η ιδανική λύση. Από την άλλη, είναι σαφής η απόφαση και άμεσα εφαρμόσιμη. Έτσι λοιπόν εσωτερικά εξετάζουμε αν πράγματι είναι απαραίτητο να υποβληθεί τροπολογία. Θα εξετάσουμε το θέμα εν ευθέτω χρόνο. Εάν αποφασίσουμε να υποβάλουμε πρόταση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τελικά θα αποφασίσουν σχετικά με τη μοίρα μιας τέτοιας πρότασης. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, δεν είναι σαφές ακόμα. Θα εξαρτηθεί από κάποιες ε, ευρύτερες ε, πολιτικές παραμέτρους για τις οποίες δεν έχω τίποτα να πω τη συγκεκριμένη στιγμή. Επίσης τέθηκε ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης από τα κράτη-μέλη, διότι η απόφαση εκδόθηκε ήδη τον Ιούνιο. Όπως όλες οι αποφάσεις ε, του δικαστηρίου που αφορούν ε, ισχύουσα νομοθεσία, ε, εφαρμόζονται άμεσα και αποτελούν αμέσως κομμάτι του κοινοτικού κεκτημένου. Γι' αυτό περιμένουμε ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αμέσως την απόφαση αυτή. Σύντομα μετά την έκδοση της απόφασης ε, συνεδρίασε η Αρμόδια Επιτροπή και θα ε, συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και θα έχουμε κατά νου το θέμα αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά τις αρμοδιότητες που έχουμε στη διάθεσή μας. Εάν είναι απαραίτητο δεν θα διστάσουμε να ξεκινήσουμε κάποια επίσημη διαδικασία Αν δούμε ότι υπάρχει παραβίαση της συγκεκριμένης διάταξης υπό το φως της πολύ σαφούς απόφασης του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ίσως η Κομισιόν ε, θα μπορεί να μας κρατήσει ενήμερους ε, σχετικά με το κατά πόσο θα εφαρμόσει τη διάταξη αυτή. Πολύ ωραία. Προχωράμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, στο σημείο 6 στην αναθεωρημένη ημερησία διάταξη. Αντιπροσωπεία ΛΥΜΠΕ στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ε, ε, τεχνολογίας πληροφορικής μεγάλης κλίμακας ε, στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Ιουλίσα, που βρίσκεται στο Ταλίν της Εστονίας. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον οργανισμό στις 29 και 30 Απριλίου. Ο νέος οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων του ΣΥΣ2, του ΒΙΣ και του Eurodac ξεκίνησε τη λειτουργία του πέρσι το Σεπτέμβριο. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις ε, εγκαταστάσεις στο Ταλίν τον Απρίλιο. Συμμετείχαν στην επίσκεψη αυτή ε, ο κύριος ε, Κοέριο και ο κύριος Λουάν και επίσης ε, στο ε, Στρασβούργο επισκέφθηκε αντιπροσωπεία ε, τις τεχνικές εγκαταστάσεις του οργανισμού αυτού. Θα δώσω τώρα λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κοέλιο να μας παρουσιάσει την έκθεση της αντιπροσωπείας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε, πήγαμε στην Εστονία και στο Στρασβούργο, στα γραφεία της Ιουλίζα, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζουμε, ε, η επίσκεψη αυτή πήρε μια διαφορετική τροπή. Κάποιες φορές η πολιτική, το πολιτικό έργο του Κοινοβουλίου αυτού δεν υποστηρίζεται όπως θα έπρεπε. Και ουσιαστικά ε, το Κοινοβούλιο έπρεπε να οργανώσει καλύτερα την επίσκεψη στο Στρασβούργο. Το κόστος δεν καλύφθηκε όπως έπρεπε και Πραγματικά αυτό είναι μια αρνητική απόχρωση στην όλη προσπάθεια. Τέλος πάντων στην Εστονία συναντηθήκαμε με τους επικεφαλείς του οργανισμού, του οργανισμού Γιουλίζα και μιλήσαμε τον, συζητήσαμε με τον ε, Υπουργό Εσωτερικών της Εστονίας. Είδαμε ότι ο οργανισμός σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπόρεσε να εκπληρώσει τις περισσότερες από τις υποχρεώσεις του και να φέρει πέρα στι αποστολέ την αποστολή που του ανατέθηκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που, ήταν, που είχε ο σήμερα ο οργανισμός να αντιμετωπίσει ήταν η έλλειψη συμμετρίας στην κάλυψη των θέσεων που έπρεπε να καλυφθούν από το προσωπικό. Πρέπει βεβαίω να υπάρχει μια σχέση βιώσιμη μεταξύ του βιωτικού επίπεδου στον χώρο του οργανισμού και τους μισθού που προσφέρονται. Όταν μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό με περισσότερους από έναν χώρους εργασία και τόπου εγκατάστασης, τότε προφανώ υπάρχουν και δυνατότητε ανισότητε. Κάποιοι κερδίζουν περισσότερα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες κάποιων που κερδίζουν λιγότερα. Στο Στρασβούργο, λόγω χάρη, περισσότερε θέσει είχαν καλυφθεί. Ενώ υπήρχαν πολλέ καινέ θέσει στην Εστονία. Διότι, όπω μπορεί κανεί να φανταστεί, για το Στρασβούργο που έχουν περισσότεροι υποψήφοι που ενδιαφέρονται παρότι για την Εστονία. Στο μέλλον ελπίζω ότι η Επιτροπή Προπολογισμών θα σκεφτεί ποιο είναι το βάρος που ένας τέτοιος συντελεστής μπορεί να έχει και στους μισθούς ώστε να μην προκαλούνται τέτοιες καταστάσεις ανισότητας. Ήταν ε, σαφές ότι η μισθολογική ε, διάσταση επηρέασε και τη διαδικασία προσλήψεων. Εδώ μιλάμε τώρα για εργαζομένους με ψηλά προσόντα και αρμοδιότητες ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων, όπως ε, για τα συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας. Δεν είναι λογικό βεβαίως ένας τεχνικός που χειρίζεται τις συστήματα, είτε είναι στο Παρίσι είτε στο Ταλίν, δεν είναι λογικός προς την πρόσληψή του να έχει τον ίδιο μισθό είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Ε, πέραν αυτού, τα πορίσματα που έχουμε σημειώσει και στην έκθεσή μας είναι να δώσουμε πράσινο φως στον οργανισμό για το έργο του και να τον συγχαρούμε για όσα έχει κάνει τονίζουμε ότι είτε στην περίπτωση της Εστονίας είτε της Γαλλίας και οι δύο χώρες στηρίζουν τον οργανισμό συγκεκριμένα διευκολύνοντας την λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς κόστος, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταβάλλει αντίτιμο ούτε επιμίσθωση για την ε, περιοχή που καταλαμβάνει ούτε στην Εστονία ούτε στη Γαλλία. Ε, κάτι που δεν ισχύει για την Αυστρία. Εκεί ε, μισθώνεται ο χώρος που καλύπτει, καταλαμβάνει ο οργανισμός ε, για τις υπηρεσίες backup. Εδώ μία σύσταση που έχουμε διατυπώσει είναι ο οργανισμός να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο καλής συνεργασίας με τα κάτι μέλη, ώστε να επωφεληθεί από την ε, πείρα των εθνικών εμπειρογνωμόνων που μπορούν ε, να, συμβάλλουν τα μάλλα στην ε, λειτουργία του ΣΥΣ 2 κατά κύριο λόγο. Ε, μεταξύ όλων των βουλευτών που επισκεφθήκαμε και την Εστονία και το Στρασβούργο νομίζω ότι παρέμεινε μια αίσθηση πολύ θετική για τον οργανισμό και μια εικόνα για το ότι είναι πραγματικά αποτελεσματικό στη λειτουργία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σίπολ θέλει το λόγο, όμως πριν τη το δώσω. Να ρωτήσω εγώ κάτι κύριε Κοέλιο για αυτό που είπατε. Εξ όσων κατάλαβα, ο οργανισμός, οι οργανισμοί μάλλον αυτοί, είναι καταναμημένοι μεταξύ των κρατών μελών και κάποιοι προσπαθούν και επιδιώκουν να έχουν ε, τα επιτελεία των οργανισμών στη χώρα τους. Επειδή μιλήσατε για την ε, διαφορετική μεταχείριση ως προς τα μισθολογικά ανάλογα με το γεωγραφικό ε, εντοπισμό των εργαζομένων, φαντάζομαι ότι αυτό διαφέρει και ως προς τις εγκαταστάσεις που προσφέρονται. Ως προς τη διαφάνεια όμως, πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να κρυφτεί το κόστος. Εσείς πώς θα το κρίνατε αυτό. Τι παρατηρήσατε. Δεν έχουμε πρόβλημα προς τη διαφάνεια. Είναι σαφές η Γαλλία προσφέρει αμυστή το χώρο το ίδιο και η Εστονία, με μια πολύ διπλωματική χειρονομία, προκειμένου να κερδίσουν την έδρα, προσφέροντας τον χώρο στον οποίο έχει κατασταθεί ο οργανισμός, δεν ισχύει αυτό για την Αυστρία. Ξέρουμε πολύ καλά το κόστος, αλλά ως προς τους μισθούς καταλαβαίνω ότι η πολιτική είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, ευρωπαϊκής κλίμακας. Δεν αφορά μόνο αυτόν τον οργανισμό. Το αν υπάρχει σχετισμός μεταξύ του επίπεδου κόστου στη χώρα και του μισθού που προσφέρεται, αυτό είναι άλλο. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι σωστή πολιτική επιλογή, διότι αν μιλούμε για υψηλόβαθμου υψηλόβαθμους τεχνικούς με μεγάλη εκπαίδευση οι οποίοι όμως δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε, μια, σε έναν διαγωνισμό. Πρόσκληση δήλωση ενδιαφέροντος δηλαδή. Ναι, το call for tender στα αγγλικά. Σε ευχαριστώ Αντουάν. Διότι προτιμούν να διατηρήσουν την σταθερότητα που έχουν εξασφαλίσει σε άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Να σας δώσω το παράδειγμα που μας δώσανε και σε εμά κάποιοι ήδη εργάζονταν σε αυτό το τομέα στι Βρυξέλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπέβαλαν καν τα χαρτιά του στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο στην Εστονία για να μην ε, χάσουν χρήματα. Και σε κάποιες περιπτώσεις ε, μας είπε ο οργανισμός ότι αρνη, υποχρεώθηκε να απορρίψει υποψηφίου, διότι ήταν πρόθυμοι υποψήφοι να επιδιώξουν το μισθό, αλλά δεν είχαν το απαραίτητο επίπεδο εκπαίδευση. Καταλαβαίνω ότι ο συσχετισμός μεταξύ μισθολογικού επίπεδου και τοποθεσίας ισχύει στην πράξη, όμως θα πρότεινα στην Επιτροπή Προπολογισμών να μελετήσει κατά πόσο σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι επιζήμιο το υψηλό επίπεδο μάλλον των μεγάλων αριθμών προσλήψεων με χαμηλότερους μισθούς. Μήπως θα έπρεπε να μειώσουμε αυτό τον ε, συντελεστή. Αλλά δεν μπορώ να το αποφασίσω αυτή τη δική μας επιτροπή. Κάποια άλλη θα το κάνει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σίπχολ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοέλιο έφυξε ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα δεν ισχύει μόνο για την Ιουλίζα. Το βλέπουμε στον τομέα της ε, ασφάλειας ε, της τεχνολογίας της πληροφορικής, ε, γενικά στον τομέα αστυνομίας και δικαιοσύνης. Οι, πραγματικά κατάλληλοι υποψήφοι να μην θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, διότι πληρώνονται καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής. Ο κύριος ε, Κοέλιο ανέφερε ότι δεν ε, μειώνει κανείς ε, τα κριτήρια, αλλά αυτό σημαίνει ότι λείπει προσωπικό. Και έτσι διακυβεύεται η λειτουργία των οργανισμών αυτών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω Στο πλαίσιο αυτών ε, των μεγάλων ε, συστημάτων συλλογής ε, δεδομένων, αναφέρθηκε το ΣΥΣ2, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν πράγματι Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν δεν είναι ασφαλής η διαφύλαξη των στοιχείων. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, ιδιαίτερα υπό το φως ε, της ε, παρούσα κατάστασης. Ευχαριστώ. Κύριε Κοέλιο, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει βρεθεί ούτε ένα πρόβλημα όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο. Ειλικρινά, οι δύο περιπτώσεις που γνωρίζω εγώ οι δύο περιπτώσεις ε, ε, διαρροής στοιχείων ε, είχε να κάνει με έλλειψη ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο λοιπόν διέρευσαν τα στοιχεία. Εμείς λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει για να αξιολογήσουμε εάν η διασύνδεση των κρατών μελών με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο είναι αρκετά ασφαλής ε, θα πρέπει να ρωτάμε τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να ε, κατηγορήσουμε ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, ούτε αυτόν τον νέο οργανισμό, διότι λειτουργεί πολύ καλά. Υπό τη δική μας αρμοδιότητα δηλαδή δεν είχαμε ούτε μία περίπτωση ε, όπου να μην ήταν ασφαλή τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω από τη Γραμματεία υπάρχει μια επιστολή προς την Κομισιόν πάνω στο θέμα αυτό για το SIS. Ελπίζω αυτό να είναι χρήσιμο. Υπάρχει κανείς άλλος που ε, θέλει να πάρει το λόγο. Στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις. Ε, αυτό είναι πολύ θετικό. Κύριε Κοέλιο, ε, είμαστε ευγνώμονες. Ε, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνατε για την Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, έχουμε άλλο ένα θέμα που θα συζητήσουμε στις 4 και 4. Δεν έχουμε συμμετέχοντες. Είναι μια ήσυχη Δευτέρα απόγευμα. Δεν με εκπλήσει που δεν είναι κανείς παρόν από τη Γερμανία, αλλά, εν πάση νομίζω ότι θα πρέπει να διακόψουμε για λίγο και να επανέλθουμε στις 4 και 4 για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη όσου έχουν δουλειά μετά από αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. 4 και 4 λοιπόν θα επανέλθουμε. Ladies and gentlemen, welcome back from your... Κυρίες και κύριοι, καλώς επιστρέψατε από το διάλειμμα αυτό αναψυχής. Να περάσουμε στο σημείο 4. Καλώς ήρθατε όσοι επιστρέψατε απλώς και όσοι έρχεστε πρώτη φορά απόψε, σήμερα το απόγευμα. Προστασία λοιπόν του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2383 JAI του Συμβουλίου. Η εισηγήτριά μας είναι η Ανθέα Μάκεντάιρ και να πω στους συναδελφούς ότι στις 19 Ιουνίου Επιτροπή λίμπε άκουσε την κυρία Μάκεντάιρ στην παρουσίασή της για την γνωμοδότηση αυτή και από τότε υποβλήθηκαν 57 τροπολογίες σε αντίθεση με κάποιες χιλιάδες που υποβάλλονται για άλλα θέματα εδώ και πριν δώσω το λόγο στην ε, μάλλον αφού δώσω το λόγο στην συγκήτρια θα προσκαλέσω τους σκιώδες που παραστάνται να παρέμβουν και όσα μέλη το επιθυμούν. Και μετά θα ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει, αν έχει την ευγενική καλοσύνη να σχολιάσει τη συζήτηση και τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Κατά πρώτον λοιπόν η κυρία Μάκαντάιρ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η έκθεση αυτή έχει να κάνει με μια απόφαση να συγκυριστούν οι ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση της παραχάραξης των νομισμάτων γενικά. Η παραχάραξη του ευρώ φυσικά είναι απειλή για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και οι σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα είναι πολύ σημαντική πτυχή της παραχάραξης. Όπως είπε ο Πρόεδρος, ήδη Είχαμε συζήτηση πάνω στο πρώτο σχέδιο της έκθεσής μου και γενικά νομίζω ότι η πρόταση αυτή ε, ότι την ε, ε, πρόταση αυτή αξίζει να την καλωσορίσουμε, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις. Καταρχήν όσον αφορά το κριτήριο της εδαφικότητας. Ήδη έχω υποβάλει τροπολογία που λέει ότι το κράτος μέλος ε, θα πρέπει να καθορίζει, θα πρέπει μάλλον να είναι το πρώτο κριτήριο κατά τον καθαρισμό της δικαιοδοσίας. Δεν νομίζω ότι ε, θα έχουν θυγεί πολύ από αυτή την τροπολογία και το άλλο έχει να κάνει με τις ελάχιστες ποινές. Η Κομισιόν θεωρεί ότι χρειάζεται εναρμονισμένη προσέγγιση ε, για να είναι αποτρεπτική. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός των κρατών μελών θεωρούν ότι τέτοιες ελάχιστες κυρώσεις ε, θα ήταν ε, θέμα υπερβολικά φιλόδοξο και ότι αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας. Επίσης, λόγω των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, η δημιουργία εναρμονισμένου συστήματος ποινών θα οδηγήσει ε, σε πολύ ε, σε μεγάλες διαφορές όσον αφορά την αποτρεπτικότητα του μέτρου και γι' αυτό θα είναι ε, μη επικοδομητική μια τέτοια προσέγγιση. Κάποιες από τις τροπολογίες μου επικεντρώνονται στις ελάχιστες ποινές και σημαντικός αριθμός φαίνεται να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Είμαι ευγνώμων προς την κυρία Σκρίφλε, Ντεγιόγκ και ε, Ταβάρης για τις τροπολογίες τους και επίσης ε, είμαι ευγνώμων προς ε, την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Φως για τις ε, τροπολογίες τους για τα εκτιμώντας. Οι τροπολογίες της κυρίας Φαγιών μου δημιουργούν κάποια προβλήματα, κάποιες από αυτές, αλλά πρέπει να πω ότι οι τροπολογίες 39 και 57 ε, είναι πολύ καλές. Για άλλες τροπολογίες έχω ερωτήσεις και νομίζω ότι αντί να σχολιάσω ε, περαιτέρω, καλό θα είναι να τα ε, ρυθμίσουμε αυτά σε συνεδρίαση των ε, σχεδόν εισηγητών. Ναι. Είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε ε, θετικό τρόπο να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία και βοήθεια των σχεδόν εισηγητών. Η κυρία Βίκστρομ επίσης με υποστήριξε πολύ στις εργασίες αυτές και προσβλέπω σε μια συνάντηση των σχεδόν για να πετύχουμε μια καλή συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η κυρία Στρίφλερ καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά τι διάφορε μελέτε αντικτύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεπίστωσε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εγκρίνει αποκλίνοντε κανόνε για να καταπολεμήσουν την παραχάραξη του ευρώ και αυτέ οι αποκλήσει αφορούν κυρίω το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων που εφαρμόζονται κατά τη παραχάραξη. Η νέα οδηγία, όπω προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπαθεί να επιβάλλει ένα, μήνυμα, ένα ελάχιστο επίπεδο κυρώσεων για όλα τα κράτη-μέλη, προβλέποντα κυρώσεις που έχουν να κάνουν με ένα εξάμεινο ή οκτώ χρόνια φυλάκισης για τα πλέον σοβαρά αδικήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και την κυκλοφορία των παραχαραγμένων νομισμάτων. Οι διατάξει αυτέ ε, διαπιστώθηκε ότι είναι αναγκαίε επειδή κράτη, κάποια δεν έχουν παρά μόνο μία ελάχιστη ποινή για το αδίκημα τη παραχάραξη, κάτι που επιτρέπει την ε, κατάσταση των παθακρακτών σε κρατημέλη ε, με την ε, λεγόμενη άγρα δικαιοδοσία ε, σε κρατημέλη που η νομοθεσία του είναι πιο ήπια. Έχουμε υποβάλει μια σειρά από τροπολογίε για την πρόταση τη Επιτροπή, η οποία στο, οι οποίε στόχο έχουν βεβαίω να παραμείνουν οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή για τι κυρώσει ανάλογα με το σοβαρό τη κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να προβλέψουν και άλλη ποινή πέραν τη φυλάκιση. Δεύτερον, τα δικήματα ή παραβιάσει που ε, είναι ιδιαίτερα σοβαρέ θα πρέπει να μπορούν ε, να υπόκεινται σε ποινή 6 μήνε το λιγότερο και μέγιστη ποινή 8 έτη. Ε, με την διάθεση να παραμείνουν οι ποινικέ κυρώσει σχετισμένε με τον παραχάραξη των νομίσματο και το εύρο τη κυκλοφορία των παραχαραγμένων νομισμάτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να καταργήσει το όριο, δηλαδή τα χρηματικά ποσά που καθορίζουν το, τη σοβαρότητα τη παραβίαση, όμω τα ποσά δεν είναι ίσω το πιο αξιόπιστο στοιχείο. Υπάρχουν σοβαρέ ανισότητε μεταξύ των κρατών ε, μελών. 6.000 ευρώ είναι ένα ποσό διαφορετικό για τα πλουσιότερα κράτη και τα λιγότερο πλούσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αφήνεται στη διακριτική ευκαιρία του Εθνικού Δικαστή. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με του συναδέλφου για να ε, προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και να βρούμε λύση σε όλα τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, now... Ευχαριστούμε. Κύριε Φαγιόν, ευχαριστώ την εισηγήτρια και σας πρόεδρε. Θα περάσω στα σλοβενικά. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ για το έργο σας και για την έκθεση που μας παρουσιάσετε σήμερα εδώ. Θα πρέπει να συζητήσουμε τι τοπολογίε που υποβλήθηκαν, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ήταν καλή διατύπωση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω αποβάλει 10 τροπολογίες ε, και οι σημερινέ συζητήσει σε ό,τι αφορά την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη ε, έρχεται σε μια στιγμή πολύ κατάλληλη λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που ακόμα βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές πολλές μάλλον ευκαιρίε για τους παραχαράκτες για να, να λάβουν δράση. Οποιοδήποτε λοιπόν μέτρο για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας είναι καλοδεχούμενο. Να πω ότι καλό θα ήταν να δούμε το θέμα των ελάχιστων ποινών. Είναι ένα σημείο στο οποίο περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο μέλλον κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και με ε, τις πολιτικές ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο. Ποιο είναι όμως το ζήτημα, ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφωνίες και πολύ διαφορετικές ποινές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι όντως ε, προχωρούν σε άγρα δικαιοδοσίας οι παρανομούντες. Γι' αυτό θα πρέπει να τους αποθαρρύνουμε με την επιβολή σοβαρών ε, ελάχιστων ποινών. Στη χώρα μου, τη Σλοβενία, ήδη υπάρχει ελάχιστη ποινή εξάμενης φυλάκισης για την παραχαράξη. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό στις συζητήσεις μας Άλλωστε δεν έχουμε συζητήσει το ευρύτερο θέμα των ελάχιστων ποινών και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, ελπίζω σύντομα, διότι έχουμε πολλά παρόμοια ντοσχέ που αυτό το θέμα ανακύπτει διαρκώς. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα έδαφο συνεννόησης εδώ με την ε, εισηγήτρια και ελπίζω αυτό να συμβεί και στις ε, διαπραγματεύσει μα από το Συμβούλιο. Ελπίζω να εγκριθεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια ώστε να συντομότερα. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίκστρομ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επικροτώ την έκθεση αυτή. Βρίσκω την ε, γραμμή της εισηγήτριας πολύ σοφή και συμμερίζομαι την άποψή της και άλλων συναδέρφων ότι δεν θα πρέπει να εισάγουμε ελάχιστε ποινές ε, σε αυτήν την πρόταση. Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν ελάχιστες ποινές στα συστήματα ποινικών κυρώσεων και θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της ε, δικαστικής ανεξαρτησίας ε, και αναλογικότητας. Κάτι τέτοιο λοιπόν ε, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που να αντίκειται στα συστήματα του ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή θέση με την καθοδήγηση της εξαιρετικής εισηγήτριάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Ταβάρη στην κυρία Ιόν εδώ σήμερα το απόγευμα. Η κυρία Ματιού, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, θα σας διαβάσω μια ομιλία που προέβλεπε να διαβάσει ο Αξελφός, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί και ζητά συγγνώμη. Υπέβαλα τροπολογίες κατά, τη ε, κατά της θέσπισης ελάχιστων και μέγιστων ποινών. Όχι γιατί δεν χρειάζεται να αρμόνιση των ποινών, αλλά θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την άγρα δικαιοδοσία και να επιδιώξουμε του στόχου τη οδηγία. Κατά κύριο λόγο, επέβαλα αυτέ τι τροπολογίε για να προκαλέσω συζήτηση. Συζήτηση, γιατί έχω την εντύπωση ότι η εναρμόνιση των ε, δικαστικών ποινών μπορεί να προκαλέσει λειτουργία στα εθνικά ποινικά συστήματα. Ο στόχο μου δεν είναι να επιβληθούν αυτέ τι τροπολογίε ε, πάση θυσία, αλλά είναι μια στρατηγική που σκοπό έχει να δούμε το ποσό των ε, ζημιών και ανάλογα να προτείνονται και ακυρώσει. Δηλαδή να επιβάλλονται ανάλογα με το σφάλμα και με το αδίκημα. Ένα παράδειγμα στη Γερμανία. Υπάρχει μια απλή κλοπή όταν κανείς ε, κλέβει κάτι, αλλά είναι διαφορετικό το αδίκημα όταν κάποιος εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός προσώπου, έχει βίαιη συμπεριφορά ή παραβιάζει έναν ε, χώρο κάποιου κτηρίου εδώ θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει να κρίνεται το βάρος του αντικείμενος ανάλογα και με το ποσό που ε, είναι το αντικείμενο της κλοπής. Δηλαδή αν κάποιος κλέψει το πορτοφόλι μιας κυρίας στο δρόμο και το πορτοφόλι έχει 5 ευρώ το αδίκημα είναι λιγότερο ε, σοβαρό σε αντίθεση με την κλοπή μιας σύνταξης 500 ευρώ. Αυτό ε, πραγματικά αντίκειται στην γερμανική λόγου χάρη αντίληψη του δικαίου στη Γερμανία. Λαμβάνεται υπόψη η χρήση όπλου ή όχι, η συνάσπιση, ο συνασπισμός σε συμμορία και ο τρόπος ε, υλοποίησης του αδικήματος. Υπάρχει λοιπόν τρόπος να βρούμε ένα κοινό συντελεστή για τα ειδικήματα. Θα πρέπει να ξεχάσουμε λίγο την έννοια των ελάχιστων και μέγιστων ποινών και να ασχοληθούμε με τις διαφορετικές εκτελέσεις του δικαίου στις διάφορες χώρες και να δούμε αν μπορούμε να αποτιμήσουμε διαφορετικά τα δικήματα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι ε, ε, στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το αποφασίσει αυτό. Διότι η ομάδα επαφής για το ποινικό δίκαιο την Τενίντε Γιόγκ μπορεί να διαματίσει εδώ σημαντικό ρόλο. Τέλος της ε, παρέμβασης του κυρίου Φως. Εδώ συνάδελφοι να σας πω και εγώ ότι όντως στο επίπεδο της πολιτικής μας ομάδας δεν έχουμε θέσει το θέμα με σαφήνεια για τις ελάχιστες και μέγιστες ποινές ή την αναρμόνιση των ποινών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως όμως είπαν κάποιοι συνάδελφοι και εδώ σήμερα, θα πρέπει ίσως να μην ανταράξουμε περισσότερο τις ποινικέ παραδόσεις και συνήθειες των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Η ιδέα αυτή δεν έχει εγκαταληφθεί. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι που στο Συμβούλιο ζητούν εναρμόνιση σε αυτό το θέμα. Ακόμη και Εάν ε, περάσαμε 18 μήνες στην Επιτροπή Κριμ με την ε, κυρία Φαγιόν, με εσάς πρόεδρε, που βλέπουμε ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, αλλά είναι δύσκολο να υπάρχει αυτή η δικαστική μετάβαση. Στο επίπεδο λοιπόν της πολιτικής μας ομάδας δεν υπάρχει κάποια σαφής τοποθέτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από την κυρία Μάκιντάιρ να απαντήσει σε κάποιες από τις παρατηρήσεις αυτές. Νομίζω ότι οι παρατηρήσει σα, κυρία Ματιό, ήταν πολύ σημαντικέ. Ε, Επίση, ε, είναι παρόν ο κύριο Τιγιόν, που είναι σκιώδη εισηγητή. Ε, θα θέλατε να πάρετε το λόγο. Τιγιον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που άργησα. Δεν ήταν πρόθεσή μου να αργήσω, αλλά συμμετείχα σε σημαντική συνάντηση στην πατρίδα μου και γι' αυτό ε, κατέφτασα στις Βρυξέλλες αργότερα από ό,τι σκόπευα. Θα ήθελα να περιοριστώ σε ένα θέμα. Έχω υποβάλει αρκετές τροπολογίες, αλλά το θέμα που έθιξε ο κύριος Φως μέσα της κυρίας Ματιού είναι πολύ σημαντικό. Είναι ζωτική σημασία στο θέμα αυτό. Και έχει να κάνει με τις ελάχιστες ή μέγιστες ποινές. Μέχρι τώρα η παράδοση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν σε ε, μέσα ποινικού δικαίου να ε, έχουμε ελάχιστε μέγιστε ποινέ, δηλαδή τα κράτη-μέλη διασφαλίζουν η μέγιστη ποινή που να μπορεί να επιβληθεί να είναι τουλάχιστον ε, ενός ε, συγκεκριμένου επίπεδου, ε, αλλά αυτό διαφέρει πολύ από τις ελάχιστες ποινές, διότι η παράδοση των κρατών μελών διαφέρει πολύ στο θέμα αυτό. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εισάγει ελαχιστε ποινες ποινέ, ενώ άλλα κράτη-μέλη όχι και στα άλλα κράτη-μέλη εναπόκειται στον δικαστή να αποφασίσει το ύψος της μηνής, να λάβει υπόψη του ελαφρυντικά ε, στοιχεία κλπ. Ε, είναι λοιπόν ε, πολύ βασική η συζήτηση αυτή και όπως είπε και ο κύριος Φως, θα πρέπει να χειριστούμε το θέμα αυτό οριζόντια. Θα πρέπει να υπάρχει μία ομάδα επαφής για το ποινικό δίκαιο. Βέβαια ε, είναι άτυπος ο διάλογος που γίνεται εκεί, αλλά υπάρχει διαφορά στο πώς ε, το βλέπουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να χειριστούμε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με οριζόντιο τρόπο και θα προτιμούσα η Κομισιόν σε μια ανακοίνωσή της ή σε κάποιο ε, έγγραφο συλλογισμού να παρουσιάσει την οπτική της για το θέμα των ελάχιστων ποινών. Ε, κατόπιν θα μπορούσε να ακολουθήσει συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για το αν μας αρέσει ε, αυτή η προσέγγιση και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κάτι τέτοιο μπορεί να σκεφτούν αν θέλουν να το εισάγουν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Δεύτερον, αν συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ελάχιστες ποινές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, θα πρέπει να ε, δεχτούμε και τη λογική συνέπεια. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα εγκλήματα που θεωρούμε τα χειρότερα. Ε, και νομίζω ότι είναι κακό πράγμα η παραχάραξη του ευρώ, αλλά νομίζω ότι η εμπορία ανθρώπων είναι χειρότερο, διότι ε, είναι κάτι που προσβάλλει την ε, σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων, που διακυβεύει την σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων. Η καλή διαδικασία λοιπόν όσον αφορά το ποινικό δίκαιο ξεκινάει με μια οριζόντια συζήτηση και θα πρέπει το χρονοδιάγραμμα αυτό να ξεκινάει με τα χειρότερα εγκλήματα. Η Κομισιόν λοιπόν ε, εισάγει τέτοια στοιχεία εδώ και εκεί. Λένε ότι ε, τα δημοσιονομικά της Ένωσης είναι υψής της σημασίας και γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, ελάχιστες ποινές σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτά είναι τα χειρότερα εγκλήματα στον κόσμο τούτον και γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογίες για να διαγράψουμε την αναφορά στις ελάχιστες ποινές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω εάν θέλει να πάρει το λόγο η Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, uh, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εκπρόσωποι της Όλαφ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε τώρα για το θέμα αυτό και για την εξαιρετική συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Επίσης να ευχαριστήσω για την άνοιξη συνεργασία και με την Προεδρία ε, του Συμβουλίου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτή την οδηγία βάσει του άρθρου 83 της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά πρώτον, για να εξυγχρονίσει το υπάρχον πλαίσιο έπειτα θελήσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ενταθεί η αποθάρρυνση, η αποτροπή της παραχάραξης κατά κύριο λόγο του ευρώ, αλλά η πρόταση μας καλύπτει και άλλα νομίσματα, βάσει της σύμβασης της Γενέβης, να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Γιατί υπήρξε αυτή η ανάγκη ε, ε, ένταση της προστασίας των νομισμάτων μας, ιδίω του ευρώ. Διότι λαμβάνουμε συνεχώς ειδήσει για το επίπεδο απειλής από την Europol με τις εκθέσεις οκτά και πρόσφατα λάβαμε και στατιστικά στοιχεία από την ECP όπου αναφέρεται και διαπιστώνεται τάση η οποία έχει πλέον αποκρισταλωθεί για πολλαπλές προσπάθειες παραχάραξης που αυξάνονται συνέχεια και μάλιστα ραγδαία. Εν της εισαγωγής των νέων ε, χαρτονομισμάτων υπάρχει ανάγκη πλέον να ε, ληφθούν κάποια μέτρα. Έχουμε προβλέψει ελάχιστες ε, ποινές στην πρότασή μας για να καλύψουμε και τις ανάγκες της αρχής της επικουρικότητας. Γι' αυτό μιλήσαμε για τις δημοσιονομικές απειλές για να δούμε τι γίνεται με συγκεκριμένε περιπτώσεις και το κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά στοιχεία. Επίσης, έχουμε χρησιμοποιήσει στατιστικά στοιχεία για να έχουμε και αριθμούς και να δούμε ποια είναι η πλειοψηφία των κρατών μελών που έχουν ή δεν έχουν εναρμονιστεί με διεθνείς κανόνες, ε, υιοθετώντας ελάχιστες ποινές για αυτή την πολύ σημαντική παραβίαση, το σημαντικό αδίκημα μάλλον παραχαραξής νομισμάτων. Κάτι που είναι ιδιαίτερα επιζήμιο και για τα θύματα αλλά και για τα κράτη. Γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει όσους συμφωνούν με την εισαγωγή των ελάχιστων ποινών στην πρότασή μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που λάβαμε αυτή την στήριξη και επίσης με ιδιαίτερη χαρά Θα συνεχίσουμε να έχουμε υποστήριξη για τις ελάχιστες ποινές ε, και στην, ε, στο φάσμα των 8 ετών. Αυτή η πρόταση υπάρχει στην, ε, στο κείμενο που υπέβαλε η Επιτροπή και θα θέλαμε να μην καταργηθεί κάτι που ήδη έχει επιβληθεί ως εκδημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αρχίσει να υλοποιείται και από τα κάτι μέλη με μια καλή μεταφορά της οδηγίας στα μέγιστα όρια. Πιστεύουμε ότι αυτό θα καλό να παραμείνει μέρος του κεκτημένου ως προς τα χρηματικά ποσά ως ανώτατα όρια ε, Ευχαριστώ να συζητήσουμε μαζί σα για να βρούμε δεύτερε απαντήσει. Καταλαβαίνουμε ότι οποιοδήποτε ε, σύστημα ποινών θα πρέπει να είναι αναλογικό ε, και δίκαιο. Να λαμβάνει υπόψη τι ελαφρυντικέ ε, συνθήκε κάποιων υποθέσεων. Γι' αυτό τόσο πολύ υπολογίζουμε στην κρίση και τη διακριτική ευχαίρεια των δικαστών που θα κρίνουν αναπερίπτωση. για να δει ο κάθε δικαστή, τι ειδικέ συνθήκες μπορεί να ισχύουν σε μια υπόθεση. Υπάρχει και μια αιτιολογική σκέψη για να καλυφθεί το σημείο αυτό. Και ένα τελευταίο θέμα. Η συγγήτρια νομίζω ανέφερε ανησυχία τις, τις ανησυχίες της για την δικαιοδοσία και την άγρα δικαιοδοσία. και εδώ ακολουθήσαμε τη ισχύοντα περί δικαιοδοσίας βάσει της απόφασης πλαισίου και στην ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχει επεφρασμένη η αρχή να ασχολείται η δικαιοδοσία κατά πρώτο λόγο με τους, ε, ε, με τους ε, υπηκόους της, τους, της κάθε χώρας. Αυτό είναι κάτι που ακόμα όμως είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε και ευχαρίστως να διαπραγματευτούμε μαζί σας για να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις στα επιμέρους προβλήματα που αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτρια για να κλείσει και να απαντήσει ενδεχομένως σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, ε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η προστασία δεν αναφέρεται μόνο στο ευρώ αλλά και σε άλλα νομίσματα. Ίσως θέλει να απαντήσει και σε αυτό. Ε, ε κυρία Μάκιντάιρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική συζήτηση σήμερα το απόγευμα και είμαι ευγνώμων προς όλους τους κοιόδης εισηγητές ε, που ε, συμμετείχαν. Είναι πολύ σημαντικό το ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η παραχάραξη οποιοδήποτε νομίσματος θα πρέπει να θεωρείται σημαντικό έγκλημα. Και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα αφορούν την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη. Εγώ λοιπόν που προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο χαίρομαι πολύ που ε, θα προστατεύεται και η Λύρα, η Βρετανική. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε να βλέπουμε δίωξη του εγκλήματος αυτού σε όλες τις χώρες. Ε, υπάρχει λοιπόν συμφωνία όσον αφορά τη σημασία των μέτρων αυτών και όσον αφορά την σοβαρότητα της παραχάραξης ε, ως έγκλημα. Ο τομέας όπου φαίνεται να υπάρχει κάποια ε, διαφωνία είναι το θέμα των ελάχιστων ποινών. Και ε, ενθαρρύνθηκα από ε, την, την υποστήριξη Μάλλον τη μη υποστήριξη για ελάχιστε ποινέ. Είχαμε κάποιε διαφωνίε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κρίμα εάν δεν προοδεύαμε στο θέμα αυτό λόγω ε, της τυχής των ελάχιστων ποινών. Ε, θα λάβω υπόψη μου λοιπόν όλες τις παρατηρήσεις που άκουσα σήμερα. Θα εκπονήσω κάποιες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και θα οργανώσω πολύ σύντομα μια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να δούμε αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε συμφωνία σύντομα. Σας Ευχαριστώ πολύ με το δικό σας όνομα και το δικό μου Κέρκοπ, που και οι δύο, θα πρέπει να περιλαμβάνει, ελπίζω, η ρύθμιση όχι μόνο το αγγλικό νόμισμα αλλά και το σκοτσέζικο. Ευχαριστώ λοιπόν. Η ψηφοφορία, ξέρετε, για το συγκεκριμένο θέμα έχει αναβληθεί και όπως είπε η συγγήτρια, θα υπάρξει μια συνάντηση των σκιωδών με την εισηγήτρια για να ρυθμιστεί το θέμα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα περνάμε στο σημείο 7. Συνθήκες εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για έρευνα, μελέτες, ανταλλαγή ε, μαθητών, κατάρτιση αμοιβόμενη ημί και ε, ο Η συγγήτρια η Σεσίλια Βίξτρομ. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ της 9 Ιουλίου η κυρία Βίξτρομ παρουσίασε την έκθεσή της ε, για την πρόταση οδηγίας προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ή το 10 Σεπτεμβρίου. 128 τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Σημειώστε ότι προς το παρόν οι τροπολογίες είναι διαθέσιμες μόνο στην γλώσσα που κατετέθησαν αλλά οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία θα γίνει στη συνεδρίασή μας στις 17 Οκτωβρίου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στην Προεδρία και την Επιτροπή. Εφόσον το επιθυμούν. Και μετά θα δώσω το λόγο στα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Κυρία Βίξτρομ λοιπόν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, την πολύ σημαντική οδηγία μαζί σας σήμερα. Καλύπτει ένα σύνολο ομάδων, φοιτητές, ερευνητές από τρίτες χώρες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ανάμιξη ουσιαστικά, η συγχώνευση δύο ισχυουσών οδηγιών και προσθέτει και δύο επιπλέον κατηγορίες. Η πρόταση της Επιτροπής είναι μια καλή πρόταση και η έκθεσή μου, η οποία όπως είπατε κατετέθη πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, έχω προτείνει ορισμένες άλλαγες οι οποίες θα βελτιώσουν την περαιτέρω το κείμενο. Έχει σημασία να βελτιώσουμε την κατάσταση, να έχουμε πιο ξεκάθαρους κανόνες και να βελτιώσουμε την ικανότητα προσέλκυσης ε, νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες να έρχονται εδώ και όχι μόνο να εργαστούν αντιμετωπίζουμε ε, μια δημογραφική πρόκληση με τον γυράσκοντα πληθυσμό μας και ακόμα και αν ήμασταν ε, ελκυστική αγορά ε, για τους εργαζομένους με συγκεκριμένες ικανότητες για, αρκετό καιρό, τώρα υπάρχουν άλλες χώρες πολύ πιο ελκυστικές. Ενώ εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Έχει φτάσει η στιγμή λοιπόν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλωσορίζω τη συμπερίληψη των δύο νέων κατηγοριών. Θεωρώ επίσης θετικό το ότι οι προβλέψεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές, ότι η πρόσβαση, η δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά εργασίας των φοιτητών υπάρχει πάντα και ότι η διαδικασία διοδότησης απλουστεύεται η πρόταση να επιτρέπεται στους φοιτητές και τους ερευνητές να παραμένουν και να αναζητούν θέσεις εργασίας ή να δημιουργούν επιχειρήσεις είναι κάτι το θετικό. Θα ήθελα η παράταση αυτή να παραταθεί μέχρι και τους 18 μήνες, 6 μήνες περισσότερους από αυτούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να διευρυνθεί το έδαφος όχι μόνο σε μία ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε όλες. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις σε σχέση με την παράταση της συγκεκριμένης περίοδου. Και ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, ε, ήδη ισχύει κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Στη Γερμανία ισχύουν οι 18 μήνες για, α, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, των ερευνών κτλ. Η Γερμανία είναι η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, ο κινητήρας της Ευρώπης. Μπορεί να μην μας αρέσει που το λένε, αλλά ε, για να το κάνουν αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι το θετικό. Και πρέπει να το διευρύνουμε στο σύνολο της Ένωσης. <clears throat> Στην Ολλανδία η αντίστοιχη περίοδος είναι 12 μήνες, ενώ στη Σουηδία είναι 0 εμείς με το που τελειώνουν τις σπουδέ τους, τους αφήνουμε 10-12 μέρες για να φύγουν από τη χώρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι προβλέψεις για τα μέλη των οικογενειών των ερευνητών θα πρέπει να εφαρμοστούν επίσης και στους φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές σήμερα μπορεί να είναι πιο ηλικιωμένοι όταν ανακληρώνουν τις ε, τριτοβάθμιες σπουδές τους και τα μεταπτυχιακά τους και πολλές φορές έχουν μια οικογένεια. Εφόσον θέλουμε να τους προσελκύσουμε όλους αυτούς θα πρέπει να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Οι ρυθμίσεις για τα κράτη-μέλη να αφαιρούν τις αδειοδοτήσεις δεν πρέπει να είναι κάτι το υποχρεωτικό και θα πρέπει να είναι κάτι το εθελοντικό. Θα δώσει στα κράτη-μέλη την δυνατότητα να εξετάζουν τις προϋποθέσεις πριν από την ανέρεση μιας αδειοδότησης σχετικά με την άρνηση της αδειοδότησης για λόγους ασφαλείας, υγείας κτλ. Να προσθέσουμε εδώ ότι θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να βασίζονται ε, ε, σε συγκεκριμένες ε, συνεντεύξεις με συγκεκριμένες αποδείξεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ξέρετε ότι ήταν η προθεσμία για τις τροπολογίες, κατετέθησαν άνω των 100, 128 Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τις τροπολογίες αυτές και είμαι βεβαία ότι η συνεισφορά σας θα καταστήσει την έκθεσή μας ακόμα καλύτερη. Πολλές από τις τροπολογίες ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση και ζητούν τη συμπερίληψη και άλλων κατηγοριών όπως μαθητές σχολείων, ε, εκπαιδευτές ε, σε διαδικασίες κατάρτισης κτλ. Ξέρω ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα στο Συμβούλιο αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης και θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε στα πλαίσια του πνεύματος συνεργασίας και συνένεσης. Αρκετές τροπολογίες αφορούν θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις των εποχιακών συμβάσεων για εποχιακών εργαζομένων. Αυτά τα θέματα είναι θέματα οριζόντιας φύσης και γι' αυτό ελπίζουμε ότι μια συμφωνία στα υπόλοιπα θέματα θα βοηθήσει να προχωρήσουμε και στο θέμα των εποχιακά εργαζομένων. Αυτό αφορά επίσης και τα θέματα των <clears throat> διδάκτρων, των ποσοστώσεων, της κινητικότητας κτλ. Έχουμε αρχίσει τη διατύπωση ορισμένων ε, συμβιβαστικών τροπολογιών και θα έρθω σε επαφή με όλους όσους τις κατέθεσαν. Όπως είπα και πριν από τις διακοπές, μπροστά ένα χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ φιλόδοξο σαν κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να δώσει συγκεκριμένη εντολή το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό θα μας δώσει να κλείσουμε λοιπόν πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός στόχος και ένα σημαντικότατο επίτευγμα για το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε εδώ στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τη συγκεκριμένη οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές που είναι παρόντες. Ε, να ζητήσω πρώτα από την κυρία Κοράτσα Πίλτ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, ε, πρόταση της Επιτροπής και την ε, έκθεση της κυρίας Βίκστρομ είναι σημαντικό να ε, καταλάβουμε ότι, πρέπει, ότι η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη για να είναι ανταγωνιστική και θα πρέπει η εκπαίδευσή μας να είναι ανάλογη, θα πρέπει να γίνει ελκυστική για σπουδαστές από τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό ότι πρόκειται για οδηγία, οπότε δεν θα πρέπει να μπούμε υπερβολικά πολύ σε λεπτομέρειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποφασίσουμε δηλαδή τι είδου ε, συμβόλαια, πόσε ώρε μελέτη, πόσε ώρε ε, σπουδών, πόσε ώρε δουλειά, ε, ούτε θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερη γραφειοκρατία για τα κράτη-μέλη με διάφορε διοικητικέ διαδικασίε και απαιτήσει. Σημαντικό είναι να απλοποιήσουμε και να εναρμονίσουμε του κανόνε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου τη συνέπεια και να διευκολύνουμε την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, για συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπω υπερβολικά σε λεπτομέρειες, ε, τα χρονοδιαγράμματα για τις ε, απαντήσεις νομίζω ότι οι 16 μέρες και το δίμηνο στην πρόταση της Επιτροπής είναι εφικτό χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν, αλλαγές, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οι 30 μέρες νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης όσον αφορά το θέμα των ε, σπουδαστών και ερευνητών και η δυνατότητα να παραμείνουν μετά την ε, ολοκλήρωση του, ε, μετά το πέρασμα του χρονικού διαστήματος. Νομίζω ότι το δεκάμινο είναι σημαντική αλλαγή για πολλά κράτη-μέλη στην Σουηδία. Δεν είναι μηδενικό το χρονικό αυτό διάστημα. Καλύπτεται κανείς από το εθνικό δίκαιο και τις δυνατότητες εργασίας να στη χώρα. Δηλαδή, αν ένας φοιτητής, ένας ερευνητής έχουν μια σύμβαση εργασίας μπορούν να παραμείνουν μετά, ε, την, ε, μετά ε, αυτό του εκπνεύσει το χρονικό αυτό διάστημα. Έτσι μπορούν δηλαδή να συνεχίσουν να παραμένουν νόμιμα στη χώρα, πάντα βέβαια με βάση την αρχή ότι δεν εξαρτάται κανείς από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας και ότι μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του όσον αφορά την ε, πρόσβαση σε εργασία για τους ε, σπουδαστές. Έχω υποβάλει σχετική τροπολογία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Ε, θα πρέπει να έχουμε την αρχή οι σπουδαστές, οι φοιτητέ, να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δεν θα πρέπει όμως στην οδηγία αυτή να αποφασίσουμε πόσε ώρε θα επιτρέπεται να εργάζονται ή όχι, διότι έτσι περνάμε στα χωράφια του εργασιακού δικαίου των κρατών μελών και όλα θα πρέπει να είναι συμβατά με τα διάφορα συστήματα των διαφόρων χωρών. Και επίσης ε, θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, να διευκρινίσει το ε, εκτιμώντας 26 και το άρθρο 31 για την ίση μεταχείριση, διότι δεν είναι σαφές ποιες ομάδες δικαιούνται η ίση μεταχείριση. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό, καθότι μόλις υιοθετήσαμε την ε, οδηγία για την ε, ενιαία άδεια. Για την κινητικότητα είναι σημαντικό θέμα και αυτό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να περάσει κανεί σε άλλο κράτο μέλο. Η επανένωση οικογενειών για του σπουδαστέ, η πρόσβαση σε οικογενειακά ε, επιδόματα και επίσης θα πρέπει να συζητηθεί το ποιες ομάδες ε, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ε, μετακίνησης. Σε Σεσίλια προσβλέπω στη συζήτηση, στην περαιτέρω συζήτηση μαζί σου και με τους άλλους και συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φαγιόν, κύριε Φαγιόν, ευχαριστώ εκ μέρους της κυρίας Φαγιόν ε, τη εισηγήτρια εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία. Στην ομάδα μα οι περισσότεροι στηρίζουν την έκθεση με 17 τροπολογίε τη Τάνια, η οποία θα συζητηθούν κατά λεπτό στην ε, συνεδρία των εισηγητών. Αυτά από την πλευρά τη Τάνια για την ώρα. Yes, and I can ask uh, Mrs. Uh, και τώρα, εκ μέρου των ε, σχεδόν εισηγητών. Η κυρία Βερζιά. Ναι, για οικογενειακούς λόγους, ευχάριστους οικογενειακούς λόγους, οι συνάδελφος δεν μπορεί να είναι εδώ, ο συνάδελφος δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον, αυτό το νομοθετικό μέτρο ε, οδεύει προς την κατεύθυνση. Ε, από την πλευρά της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Παιδείας, να πω ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό και βλέπουμε ότι είναι πολύ αλλοδαπή που υπέρχονται στις χώρες μας με τέτοιους σκοπούς. Έχουμε ε, υποβάλει τροπολογίες με στόχο την απλούστευση κατά κύριο λόγο. Αλλά από αυτήν την ε, ακριβώς την οπτική γωνία υπάρχει και μεγαλύτερη δυσκολία. Καταλαβαίνω τη θέση του ΕΛΚ αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι πρέπει να προσκληθούν τα κράτη-μέλη να σεβαστούν και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο σύνολό τη. Οπότε, καλό θα πρέπει να είμαστε συνεπεί ε, στην ισορροπία που θέλουμε να εξεύρουμε μεταξύ το τι ε, βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Ω προ τα θέματα αυτά, οι τάσει των κρατών μελών βλέπουμε να μην είναι πολύ ε, κοντινέ αυτέ που θα ελπίζαμε. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ώστε να παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την νομοθεσία του. Και πραγματικά θα εκφράσω τη χαρά μου αφού συμβεί κάτι τέτοιο. Um, Ευχαριστώ. Πριν στραφώ προ την Επιτροπή, να σχολιάσω κι εγώ σαν σκιώδης της πολιτικής μου ομάδας των συντηρητικών. Οι στόχοι δεν είναι κακοί, θέλουν να βελτιώσουν ε, την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πόσο ελκυστική μπορεί να είναι για τους ε, μορφωμένους μετανάστες. Ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό πραγματικό κόσμο και σαν οικονομίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε εγκεφάλους από άλλες περιοχές για να συνεισφέρουν στις προσπάθειες που κάνουμε. Όμως, στόχος των μεμονωμένων κυβερνήσεων πολύ συχνά είναι η μείωση της μετανάστευσης. Παρ' όλα αυτά κάποιες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να προσελκύουν υψηλής ποιότητας μετανάστες, φοιτητές και ερευνητές, ιδιαίτερα για τον πανεπιστημιακό τομέα. Πολλά μέτρα λοιπόν λαμβάνονται και σε εθνικό επίπεδο και τα θέματα γενικότερα της μετανάστευσης ανήκουν στις αρμοδιότητες των κυβερνήσεων περισσότερο και των εθνικών πολιτικών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τα εξισορροπήσουμε τα πράγματα λοιπόν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίζουν τις δικές τους πολιτικές, πιστεύω. Πιστεύω όμως ότι έχει μεγάλη σημασία να έχουμε στη διάθεσή μας μια σωστή, ξεκάθαρη κατανόηση το ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση ένα άνισο, άδικο και καταχρηστικό τρόπο αντιμετώπισης αυτών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέροντας τις γνώσεις τους μαζί τους για το κοινό καλό. Λοιπόν, η πρόταση είναι μια καλή πρόταση, σημαντική πρόταση χρήζει περαιτέρω συζήτησης και περιμένω τώρα ε, και αυτά που έχει να μας πει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη δική του πλευρά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Βίξτρομ αλλά και τα μέλη του Κοινοβουλίου που κατέθεσαν τις τροπολογίες οι οποίες εν πολλής στηρίζουν την πρότασή μας, αν και μερικές φορές είναι πιο φιλόδοξες οι τροπολογίες από το δικό μας επίπεδο φιλοδοξίας. Βρισκόμαστε σε μια αρκτική θα έλεγα φάση των διαπραγματεύσεων Παρ' όλα αυτά τα πράγματα πάνε αρκετά γρήγορα και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουμε βέβαια, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το ότι πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν με την προϋπόθεση βέβαια ότι το κείμενο θα παραμείνει φιλόδοξο και ότι δεν θα υπάρξουν παλινοδίες σε σχέση με το τι έχουμε τώρα. Έχουμε ήδη δύο οδηγίες για τους ερευνητές φοιτητές και εν μέρη και για τους μαθητές και δεν θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω παρακαλώ. Ευχαριστώ λοιπόν για μια ακόμη φορά για την έκθεσή σας. Όπως είπα οι περισσότερες από τις τροπολογίες στηρίζουν την πρότασή μας και μέσω νέων κατηγοριών που πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές. Πράγματι στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα, στηρίζεται η διαδραστικότητα των πολιτικών μας, γίνεται πιο ελκυστική η ένωση στους νέους επιτρέπονται περισσότερες πολιτιστικές ανταλλαγές και προστατεύονται οι νέοι από την εκμετάλλευση ε, με καταχρηστικό τρόπο. Θέλετε να στηρίξουμε την ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να υπάρχει επίσης και η δυνατότητα στους φοιτητές και τους ερευνητές να μείνουν και μετά από τις σπουδές τους και είτε να δημιουργούν επιχειρήσεις είτε να βρίσκουν θέσεις απασχόλησης. Να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η πρόταση είναι να επιτρέψουμε στους νέους αυτούς να παραμείνουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή όμως έχουν δημιουργήσει μια επιχείρηση ή έχουν βρει μια θέση, τότε θα ισχύσει η εθνική ρύθμιση κάθε φορά. Κάνετε ένα επιπλέον βήμα σχέση με την αρχική μας πρόταση Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το ότι ήδη έχουμε ένα επίπεδο εναρμόνισης. Κατανοώ βέβαια την, τη σημασία της πρότασης που υπάρχει έτσι ώστε να αφαιρείται η αδειοδότηση, η άδεια παραμονής και τα λοιπά σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό τίθεται στο επίπεδο εθνικό στα πλαίσια της νέας κινητικότητας που εκεί ισχύουν ορισμένοι κανόνες διαφορετικοί από τους κανόνες που ισχύουν για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την άρνηση εισόδου. Πρέπει να προσθέσει αξία λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συγκεκριμένη οδηγία, πρέπει να είμαστε φιλόδεξοι και να πούμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία έτσι ώστε να συζητήσουμε και το θέμα της οδηγίας της σχετικής με την κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Υπήρξε μία συγκεκριμένη ερώτηση από πλευράς της κυρίας Μπίλτ για την αύξηση θα έλεγα. Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε για τα δικαιώματα των φοιτητών και τα ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατύπωση της συγκεκριμένης πρότασης. Ε, τα ίσα δικαιώματα τα οποία χορηγούνται μέσω της έκδοσης της άδειας παραμονής δεν αφορούν μόνο αυτούς οι οποίοι εργάζονται, αλλά και αυτούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και όλες τις άλλες κατηγορίες όπως τους φοιτητές, τους ερευνητές και συμπληρωματικά εμείς προτείνουμε να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα και να καλύψουμε και τις ανάγκες των ερευνητών. Λέμε να μην υπάρχουν περιορισμοί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για αυτούς και σχετικά με τα οικογενειακά τους δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα. Κάνουμε κάποια επιπλέον βήματα ε, τα οποία δεν υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία Προτείνουμε σαν παράδειγμα και οι φοιτητές και οι μαθητές και οι αμοιβόμενοι ερευνητές και ε, οι εργαζόμενοι ΟΠΕΡ να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε λίγο περισσότερο στο κείμενο και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα προχωρήσουμε σύντομα. Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και σε τεχνικό επίπεδο φυσικά γι' αυτό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της Λιθουανικής Προεκτείας, Προεδρίας, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να λαμβάνω το λόγο ως ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον πολύ ε, ενεργό ρόλο που ανέλαβε στην εξετάση αυτού του θέματος. με τροπολογίες που ενθαρρύνουν και το Συμβούλιο να επιταχύνει, γιατί ταχύτητα ήταν το βασικό στοιχείο της εισηγήτριας. Να προχωρήσουμε λοιπόν γρήγορα, ε, κάτι που βλέπουμε να έχει δώσει άλλωστε ως τακτική τα πρώτα αποτελέσματα με τις ε, γενικές κατευθύνσεις για τη μελλοντική τοποθέτηση του Συμβουλίου. Έχοντας λοιπόν ακούσει τη συζήτηση περί τροπολογιών, αυτές που προτείνατε εσείς, κάποιες ήταν πραγματικά τροπολογίες με τις οποίες θα μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί και εμείς τα συζητάμε, όπως ότι το κείμενο χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση και γιατί πρέπει να ορίσουμε καλύτερα την ε, έμιστη ή άμιστη κατάρτιση, το άρθρο περισσότερα στο φίλων χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση και να ευχαριστώ και την κυρία Κοράτσα Μπίλτ για την ε, παρέμβασή τη, αν προφέρω σωστά το όνομά τη, για την ανάγκη ευελιξία προκειμένου να πετύχει η εισαγωγή εργατικού ε, στα διάφορα εθνικά συστήματα. Αυτό το συζητάμε και στο Συμβούλιο. Υπάρχουν μεγάλε αποκλήσει από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε ένα μεγάλο βαθμό ευελιξία ώστε να εξυπηρετούνται όλε οι ανάγκε Πάντω να θυμίσω και το πλαίσιο του στο οποίο είναι αντικείμενο διαπομάτευση η οδηγία αυτή. αρκετά χρόνια μετά την έναξη της οικονομικής κρίσης, κάποια κράτη-μέλη έχουν τεράστιους αριθμούς ανέργων. Σε κάποια κράτη-μέλη η ανεργία των νέων αγγίζει το μισό πληθυσμό της νεολαίας, των νέων περίπου. Έτσι το Συμβούλιο ε, έχει αρχίσει να εξετάζει με σοβαρότητα το γεγονός ότι μετά την οικονομική κρίση ε, επηρεάζεται και κλειδονίζεται η αγορά εργασίας των κατεμελών. Θέλουν λοιπόν ε, τα κατεμελή να προστατεύσουν το καθένα τη δική του αγορά εργασίας. Αυτό έχει ακουστεί και στο Συμβούλιο και γι' αυτό είναι κάπως πιο διστακτικό το Συμβούλιο προς την πρόταση αυτή. Θέλει περισσότερες εγγυήσεις προκειμένου να αποφευχθούν κακοχρησίες του συστήματος, όπως θα προκύψει την οδηγία. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάθε πρωτοβουλία από το Κοινοβούλιο που είναι πιο φιλοδόξη από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει δεκτή με μεγάλη επιφυλακτικότητα από την πλευρά του Συμβουλίου. Τι άλλο συμφωνούμε ότι οι φοιτητέ, οι μαθητές και όλη αυτή η άντληση εγκεφάλων από τρίτες χώρες θα πρέπει να διευκολυνθεί γιατί η Ευρώπη τα χρειάζεται όλα αυτά. Και το Συμβούλιο εξετάζει με θετικό βλέμμα την διευκόλυνση του προγράμματος κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτό είναι σημαντικό να ξαναδούμε το πρόγραμμα για το ICT και τη σχετική οδηγία, γιατί αυτό θα μας ε, ε, χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευση και πρότυπο για να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο διακινητικότητας με το μέλιο και αυτή την οδηγία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο. Ίσως να ολοκληρώσω εδώ και απλώς να σας ευχαριστήσω ξανά για την εξαιρετική σας δουλειά και την ταχύτατη αντιμετώπιση και για Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Θα ζητήσω από την ε, εισηγήτρια να κλείσει τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Chairman, quoting yours. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έχετε πει και εσείς, ζούμε σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όπως είπαν οι συνάδελφοι, μιλάμε για ανταγωνισμό, καινοτομία και θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εξειδικευμένο ε, εργασιακό ε, δυναμικό. Και όπως είπε η συνάδελφος Κοράτσα Μπίλτ, ποτέ να μην προσθέτουμε γραφειοκρατία, αλλά να εναρμονίζουμε τους κανόνες, να ε, διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικαίου και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν τη στιγμή που έχουν φτάσει. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις θέσεις μας, να καλωσορίσουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν ήδη λάβει εξαιρετική εκπαίδευση στα πανεπιστήμια μας, να παραμείνουν, ε, να συμμετάσχουν για παράδειγμα σε ερευνητικέ ομάδες στην Ευρώπη, σε διάφορους τομείς. Όσον αφορά τη σωστή ισορροπία που θα πρέπει να βρούμε Είμαι βέβαιη ότι αυτό μπορεί να γίνει. Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο θέλει να ακολουθήσει κατά καιρούς άλλη, προσέγγι... άλλη κατεύθυνση, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα βρούμε ένα πολύ καλό πνεύμα συμβιβασμού και ότι θα καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπερβολικά πολλοί ικανοί νέοι παίρνουν διδακτορικό στα πανεπιστήμια μας και μετά φεύγουν για τις Ηνωμένε Πολιτείε, τον Καναδά και την Αυστραλία και δεν επιστρέφουν. Τους δίνουμε λοιπόν εκπαίδευση χωρίς να υποφεληθούμε ποτέ από τις ε, ικανότητές τους. Ε, αυτό θα πρέπει να το σταματήσουμε. Ε, βλέπουμε λοιπόν διαφυγή εγκεφάλων και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες ε, και θα πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά και να σταματήσει αυτή η πρακτική. Μπορεί να συζητήσει κανείς την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, εγώ έτυχε να σπουδάσω σε ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας μου ε, και ο Πρίτανης μου είπε ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να λυθούν. Οι ερευνητές ε, αυτοί μπορεί κάποια μέρα να βρίσκονται σε ομάδα έρευνας που θα λύσουν το πρόβλημα του AIDS ή άλλα σοβαρά προβλήματα. Γιατί λοιπόν να τους παρέχουμε μια εξαιρετική εκπαίδευση και κατόπιν να τους βλέπουμε να αποχωρούν από την Ήπειρό μας. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η πρόκληση. Θα πρέπει με ανοιχτό πνεύμα αλλά και αποφασιστικότητα να μην θέτουμε όρια στους εαυτούς μας, ε, να ε, μην πνιγόμαστε στη γραφειοκρατία. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό με ανοιχτό μυαλό και με προσανατολισμό το μέλλον. το μέλλον θα μας φέρει αυξημένο αριθμό προκλήσεων και με ευελιξία και ανοιχτό πνεύμα θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μία ένωση ελεύθερης κινητικότητας, ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας και ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης με καινοτομία και ανταγωνισμό. Ας είμαστε λοιπόν φιλόδοξοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή και προσλέπω στην συνέχεια της συνεργασίας μας για να εξετάσουμε την πρόταση άρθρο προς άρθρο και στο, τελικά πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά δεν ε, ολοκληρώσαμε τελείως, διότι η κυρία Παπαδοπούλου δεν ε, μπόρεσε να παρευρεθεί νωρίτερα, είναι όμως, ε, έχει συντάξει όμως ε, το σχέδιο γνωμοδότηση τη επιτροπή απασχόληση και θα ήθελε να πει λίγα λόγια. Ελπίζω να συμφωνεί η συγκήτρια. Παρακαλώ. Uh, Ζητώ συγγνώμη που δεν ήρθα νωρίτερα, αλλά έχουμε προβλήματα με τα ωράρια των αεροπλάνων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τη Σεσίλια. Είμαι βέβαια ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε βάθος γιατί πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Ε, προσπαθώ να δείξω μια κάποια ευρύτητα πνεύματος. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα. Μιλάμε για τη διαρροή των εγκεφάλων. Υπάρχει αυτό και για αυτούς οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και λόγω των οικονομικών προβλημάτων και λόγω των προβλημάτων απασχόλησης στις χώρες αυτές, οι χώρες αυτές υποφέρουν. Και οι εγκέφαλοι αυτοί δεν πηγαίνουν στη Γερμανία, στη Βρετανία ή στην Αυστραλία, προσπαθούν να βρουν θέσεις απασχόλησης στον αραβικό κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα των πολιτικών μηχανικών, των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων κτλ. Ε, βλέπω το θέμα αυτό κυρίως από πλευράς απασχόλησης και να σας πω την αλήθεια, είχα κάθε πρόθεση να ικανοποιήσω όλες τις προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην πρόταση αυτή της Επιτροπής. Όμως, Υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Και αυτό ε, γιατί όταν έρχεται κανείς από τη Σουηδία ε, ε, ή τη Γερμανία ή έστω και την Κεντρική Ευρώπη έχει διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος της διαρροής των εγκεφάλων των Ευρωπαίων. Όταν υπάρχουν κενές θέσεις απασχόλησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν ανταγωνιστικές πολιτικές από πλευράς χωρών των τρίτων ε, χωρών, για τους νέους των τρίτων χωρών, θα πρέπει να προβλέπονται αντίστοιχες τέτοιες ρυθμίσεις και για τους ε, φοιτητές που προέρχονται από τις δικές μας χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, κάποιες δυνατότητες να βοηθήσουμε να σπουδάσουν και να εξειδικευτούν οι μορφωμένοι νέοι Ευρωπαίοι και να επανέρχονται στις χώρες τους όμως για να μπορούν να ε, βοηθούν στην ανάπτυξή τους. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι όταν λέμε ότι αν βοηθήσουμε τις οικογένειες να έρθουν στην Ευρώπη τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για την Ευρώπη. Είναι πιο περίπλοκα τα θέματα, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες ήταν εθελοντικές ε, και θα έλεγα και τώρα καθίστανται υποχρεωτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο κάνει μία πρόταση η οποία δημιουργεί πάρα πολλές κατηγορίες εκπροσώπων πολιτών από τρίτες χώρες και δεν μπορούμε όλες αυτές τις κατηγορίες να τις βάλουμε στην ίδια οδηγία γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές. Συγχαίρω λοιπόν τη Σεσίλια για τη σκληρή της δουλειά. Σε κάποιες από τις θέσεις της έχουμε διαφορετικές απόψεις σε επίπεδο απασχόλησης, αλλά θα θέλαμε πάντως να πούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε σε επίπεδο ανθρωπιστικό και σε επίπεδο ίσων ευκαιριών ε, οι άνθρωποι αυτοί να μην την χάνουν εκμετάλλευσης και ταυτόχρονα να σεβόμαστε τις υπάρχουσες συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνθήκες και καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Και να μην ξεχνάμε επίσης και την αρχή της επικουρικότητας, γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν για το τι θα πρέπει να κάνουν στις χώρες τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στο τέλος της συζήτησης. Να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου. Ολοκληρώσαμε τη μερίσια μας διάταξη διότι το σημείο 8 έχει αναβληθεί. Η κυρία Μπένοβα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Ωστόσο, πρέπει να καθορίσουμε η ημερομηνία, πρέπει να καθορίσουμε προθεσμία την κατάθεση τροπολογιών για να μπορέσει να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. 24 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών το μεσημέρι. Και ε, αύριο το πρωί 9 η ώρα έχουμε το πρόγραμμα καταχώρησης ταξιδιωτών. Μπορούμε σήμερα λοιπόν να τελειώσουμε νωρίς σήμερα, να ετοιμαστούμε για αύριο το πρωί. Στο μεταξύ σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λήξη της συνεδρίασης. Ευχαριστώ.